Ε, ψηφοφορίες, έκθεση Νεγκρέσκου, η κοινοτοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Μία μόνο ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Νόβακοφ για την κινητοποίηση πάλι του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης μία μόνο ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φερνάντε σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Τροπολογία 1. Υπέρ. Για να τάσει τους χειρός παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. κτιμώντας ή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε η μονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκθεση στάες. Ορισμός μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κύριος Σάμο Γέρεμπε. Ψηφίζουμε με, ε, με μυστική ψηφοφορία. Άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκθεση Σόλτες. Ορισμός, ε, διορισμός μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κύριος Μίχαηλ Κοσλόφ. Σε πάλι μυστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Σόλτες, διορισμός μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κύριο Γιάνν Γκρέγκορ. Πάντοτε με μυστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκθεση Σόλτες για τον διορισμό μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, η κυρία Λάντισλαφ Μπάλκο. Ε, μυστική ψηφοφορία Άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διορισμός μέλος του, Ευρωπαϊ... του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρία Βοησικόφσκη. Ο κύριος Βοησικόφσκη, ε, μυστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στο ψήφισμα για την ε, ε, ένσταση στο άρθρο 106, σύμφωνα μάλλον με το άρθρο 106 του κανονισμού που αφορά την ανανέωση της έγκρισης της δραστήριας ουσίας γλυφοσάτης. Πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής ΕΝΒΗ, παράγραφος 1, τροπολογία 44, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία 9. Πάντοτε παραγραφός 1, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 10, σε 9 τμήματα. Πρώτο τμήμα, ε, διανατάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα. Ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα, Για διανατάσσεως ισχυρός υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Έβδομο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 8ο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος της Ψηφοφορία εγκρίνεται. Ένα το τμήμα. Ονομαστική κλίση άρχεται. La votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Approvato. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 καταπίπτει. Τροπολογία 11. Έχουμε μια προφορική τροπολογία του κυρίου Ντελαέ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Λειτουργεί, μάλιστα. Ωραιότητα. Κύριε Πρόεδρε. Σε πνεύμα συνεργασίας για να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σύγκληση απόψεων και να ξεπεράσουμε τις διαφορές, προτείνω την εξή τροπολογία για την παράγραφο ε, στην παράγραφο 11 ζητά από την Κομισιόν να ανανεώσει την έγκριση του Γλυφοζάτ για μια περίοδο το πολύ 7 ετών υπενθυμίζει ότι ο κανθουμός 1107 του 2007 δίνει στην Κομισιόν τη δυνατότητα να αναστείλει την έγκριση ενός προϊόντος στη διάρκεια της έγκρισης του εάν δεν εκπληρεί πλέον τα κριτήρια έγκρισης. Ευχαριστώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Υπάρχουν 40 που σηκώνονται, όχι. Ε, τότε θέτω σε ψηφοφορία την 11 που τροποποιείται σε δύο τμήματα. Σε δύο τμήματα άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Scusate, allora fermiamoci un attimo. Για σταθείτε λίγο, για σταθείτε. Ci 40 parlamentari Έχουμε 40 ευρωβουλευτές που είναι αντίθετοι. Ή δεν έχουμε. Ναι, θα έλεγα ναι. E eh, ναι, είναι 40. Μα ποιο είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι πολύ αργά, γιατί προφανώς, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, εντάξει, δεν είμαστε σε ρίγκ. Προφανώς οι συνάδελφοι που είναι αντίθετοι άκουσαν από τη μετάφραση λίγο καθυστερημένα αυτό που είπα εγώ και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν αν... Ε, αυτό πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν, την ελευθερία του να έχουν αντίρρηση. 40 λοιπόν βουλευτές ήταν. Άρα λοιπόν η προφορική ε, καταπίπτει. Περνάμε τώρα στα δύο τμήματα της τροπολογίας 11 Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Η τροπολογία 20 καταπίπτει. Η τροπολογία 46 ονομαστική κλίση. Άρχεται. La votazione chiusa. Τέλος της πληροφορίας. Respinto. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47D. Ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Διανατάσσεως της χειρός. Πιπέρα, κατά, απόχες, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Διανατάσεις της χειρός. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Δεν θέλετε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, μάλιστα. Τροπολογία 12. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Έγκρινεται. Τροπολογία 49 σε δύο τμήματα. Ε, ονομαστική κλίση. Το πρώτο τμήμα. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Διανοτάζει τους χειρός. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Τι θέλετε 37. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Διανατάσσεω της ισχυρός. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 13 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 51D. Διανατάσεις της είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 21 δυνατά στις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 15 ονομαστική κλίση άρχεται τέλος απορρίπτεται τροπολογία 16 ονομαστική κλίση άρχεται Τέλος. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας D, τροπολογία 39, D, με ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 για την εκτιμώντας D άρχεται τέλος απορρίπτεται Εκτιμώντα E. Ε, τροπολογία 40D άρχεται τέλος απορρίπτεται. Τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, πάντα με ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 σε δύο τμήματα, διανατάσεις χειρός, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τροπολογία 41 υπέρ. Τι θέλετε να επαληθεύσουμε, ας επαληθεύσουμε για το δεύτερο τμήμα, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Διανατάσσεως χειρός. Α, όχι, συγγνώμη, έχει καταπέσει. Η 41 έχει καταπέσει. Ε, εκτιμώντας όμικρον τροπολογία 5, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απέριπτε αιτιολογική σκέψη Ε, τροπολογία 42 με ονομαστική 43 ονομαστική κλίση. 42D d ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Απερίφθη, τροπολογία 6, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη Ο. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. 43D είναι η τροπολογία που ψηφίζουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίπτει. W, τροπολογία 8, με ανάταση χειρών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 18, με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 22, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Τροπολογία 23 μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 με ανάταση χειρών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. θέλετε έλεγχο για την 24 βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία ελέγχου. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 διανάταση χειρών. Υπέρ. Κατά. Αποχές αν δεν τα σηκώνετε τα χέρια σας, πού να ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 27. Διανατάσεως. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Καλά, να κάνουμε έλεγχο. 27 ψηφοφορία ελέγχου άρχεται. Εγκρίθηκε. 28 μονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 διανατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30. Έλεγχος για την 30 βεβαίως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Διανατάσσεω χειρό και πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Κάνουμε καλύτερα έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Όχι. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίκη. Περνάμε στην έκθεση Καλνιέτε, Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Θέλετε το λόγο. Μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 1, σε, τρεις, σε τρία κομμάτια. Πρώτο τμήμα με ανατεσχυρών. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. απερίφθη τρίτο τμήμα με ανάθεση χειρών υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Πάντα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Το αρχικό κείμενο σε τρία κομμάτια πάντα με ονομαστική κλίση κάθε τμήμα άρχεται για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα πάλι ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγωγος 9. Το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 σε τρία τμήμα, πάντα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έγκρινε τμήμα. Ονομαστική κλίση. Πάντα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 11 το αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12 το αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 17. Το αρχικό κείμενο με δίχως ονομαστική κλίση ανατεσχυρών πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 23. Το αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα με ανατασχηρών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 26 αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση άρχεται πέρας εγκρίνεται παράγραφος 27 το αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση άρχεται πέρας Εγκρίνεται. Παραφορ 45, τροπολογία υπαριθμών 2, ψήφι υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη σε, σε δύο τμήματα, αρχικό κείμενο υπέρ του πρώτου, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Υπότιτλος μετά από την αιτιολογική σκέψη νη, αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα του, του κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απερίφθη τελικά το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλνιέτη. Περνάμε στην έκθεση Μέσεριτς εφαρμογή και μεταρρύθμιση της στρατηγικής για την Κεντρική Ασία, παράγραφος 3, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ανατασχυρών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, έλεγχος, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 65 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διανατάσσεω τη χειρό υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 89 του αρχικού κειμένου ποιοι είναι υπέρ πρώτο τμήμα δεύτερο, ε, κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 90. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 110 το αρχικό κειμένο σε διατμήματα πρωτοτμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 149. Α, θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Για το δεύτερο τμήμα τη παραγράφου 110 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα, Απορρίπτεται. Ναι, αλλά όμως να σηκώνετε τα χέρια σας, αλλιώς θα κάνω λάθος. 149 αρχικού κειμένου, υπέρ, κατά αποχές θα λέγω ότι εγκρίνεται όμως σας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα είναι άρχεται εγκρίνεται 145 τοπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Μέσεριτς. Τώρα περνάμε στο ψήφισμα για την επιδημία του ιού Ζήκα. Πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής NV, το παράγραφος 5 μετά την παράγραφο 7, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Εντάξει, έλεγχος ηλεκτρονικός για την 5 άρχεται. Τέλος. Τροπολογία 6. Υπέρ κατά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 για το τρίτο τμήμα. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. τη χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Παράγραφος 19. τη χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19 καταπίπτει. Παράγραφος 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας U, τροπολογία 3 να τάσω της χειρός υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. E Και τώρα περνάμε στην κατάσταση στην Πολωνία. Πριν να προχωρήσουμε στο πρόταση ψηφίσματος, έχουμε μία πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας από πλευράς του κ. Καμάλ, που ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του ECR θα ήθελα να προτείνω την αναβολή του ψηφίσματος υπό τη άρθρα 185 και 190. Ο Επίτροπος Τίμερμαν μετέβη στην Πολωνία για να συνομιλήσει με την πολωνική κυβέρνηση την περισμένη εβδομάδα και ο κύριος Τίμερμαν επανήλθε από περισσότερο, ε, θα επιστρέψει λίγες μέρες για περισσότερο διάλογο και γι' αυτό λέω να αναβάλουμε μέχρι όταν να έχουν γίνει αυτές οι συναντήσεις. Σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε αυτή την κατάσταση με διάλογο περισσότερο παρά με ε, μικρότητες. Ε, το ψήφισμα, αν θέλουμε πραγματικά να επιληθεί το ζήτημα με φιλικό τρόπο, είναι προς το συμφέρον μας να προχωρήσουμε σε συνομιλίες ανάμεσα στην πολωνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά τότε ε, νομίζω πως έτσι μπορείτε να συμφωνήσετε σε αυτό το αίτημα. Να αναβληθεί μέχρι μετά τις συνομιλίες το ψήφισμα. Υπάρχει κάποιος που να είναι υπέρ, ζήτησε το λόγο η κυρία Βυζνιέσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στις 15 Ιανουαρίου ζητήσαμε από την Κομισιόν να μας δώσει τη νομική βάση της παρέμβασης της Κομισιόν στα εσωτερικά θέματα της Πολωνίας. Ζητήσαμε να μας εξηγήσει σε ποιο σημείο των συνθηκών βασίστηκε η Κομισιόν. Έχουν περάσει τρεις μήνες και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από την Κομισιόν. Ενώ η προθεσμία απάντηση για κάτι τέτοιο είναι έξι εβδομάδες. Η Κομισιόν δεν μπόρεσε να μας υποδείξει σε ποιο σημείο της συνθήκης ε, βασίζεται αυτή η παρέμβασή της γιατί δεν υπάρχει κάποια τέτοια βάση. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση στα εσωτερικά θέματα ενός κρατούς μέλους χωρίς να παραβιαστούν οι διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας ζητώ να αναβληθεί η ψηφοφορία του ψηφίσματος μέχρι ό,τι η Κομισιό μας αναφέρει τη νομική βάση. Ο ιατρός θα πρέπει να θεραπεύσει τον εαυτό του. Θέλετε να αλλάξετε την νομοθεσία στην Πολωνία, αλλά παραβιάζετε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Φύγοντα στην Πολωνία, θίγετε την Ευρώπη. Ήσασταν σαφέστατοι. Υπάρχει, ήσασταν σαφέστατα υπέρ της πρότασης του κ. Καμάλ. Θέλει κανείς να ψηφίσει κατά αυτής της πρότασης ο κ. Πιτέλα. Παρακαλώ. ήθελα ταπεινά να θυμίσω σε ολόκληρη το σώμα ότι μια χώρα είναι ελεύθερη να εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν μπορεί να την αναγκάσει. Το επιλέγουν οι ίδιοι οι πολίτες. Αλλά τη στιγμή που προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, καμία παρέμβαση, καμία παρέμβαση, αλλά νόμιμο και ε, ενδιαφέρον και ε, καθήκον από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δει τι συμβαίνει στην ίδια της την οικογένεια γιατί η Πολωνία είναι η οικογένειά μας και εμείς ενδιαφερόμαστε για την τύχη των Πολωνών πολιτών αυτό το ψήφισμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια των αποτελεσμάτων της σύμβασης της Βενετίας που σαφώς ε, ε, μίλησε και θέλουμε να γίνει σεβαστή στο μάλλον το συμφέρον του λαού της Πολωνίας. Ευχαριστώ κύριε Πιτέλα και τώρα ψηφίζουμε για την πρόταση αναβολής όπως πρότεινε ο κύριος Καμάλ. Με ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Περνάμε στο πρόταση ψηφίσματος των πέντε πολιτικών ομάδων, παράγραφος 10, τροπολογία 3, ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές. Ε, ε, μία επαλήθευση κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική κρίση. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 στο εκτιμώντας π. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ε, απορρίπτεται. Μετά από το εκτιμώντας π, τροπολογία 2, ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται. La votazione è chiusa. Approvata. E Εγκρίνεται. Terminano qui, no? Sì, sono le dichiarazioni di voto. Sì. Allora, terminano qui le votazioni. Εδώ τελειώνουν λοιπόν οι ψηφοφορίες και περνάμε τώρα στις δηλώσεις, επεξηγήσεις μάλλον ψήφου. Θα περιμένω κάποια στιγμές για να βγουν οι συνάδελφοι από την αίθουσα.